ότι η Επιτροπή μας στην κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση και μυστική ψηφοφορία να εγκρίνει την υποψηφιότητα του κυρίου Βέσπερκ για τη θέση του μέλους του Ελεκτικού Συνεδρίου. Πέρασε επιτυχώς λοιπόν ο υποψήφιο. και θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξης προβλέπει την εντολή για τον τριμερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού του 2012. Ο εισηγητής τη έκθεση είναι ο κύριο Χατζημαρκάκης και θα υποβάλει κάποια σχόλια. Έχετε το λόγο, κύριε Χατζημαρκάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι η τροπολογία υπαριθμών 8 του κυρίου Κοτσολίνο ε, αποσύρθηκε. Και επίσης ε, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στο 10, στην τροπολογία 10. Κοιτάξτε, εάν η τροπολογία υπαριθμών 9 και συγκεκριμένα μόνο το πρώτο κομμάτι της εγκριθεί, ε, πρόκειται για την τροπολογία του κυρίου Καταλίν Ήβαν. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει και η τροπολογία υπαριθμών 10. Τουλάχιστον έτσι το κατάλαβα. Ε, βλέπω τη γραμματεία που νεύει καταφατικά. Απλά ήθελα να σε για αυτές τις δύο αλλαγές. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο κύριος καία Εμείς ε, στην ομάδα, εργασία μας, ε, ομάδα εργασίας αποφασίσαμε την τροπολογία υπαριθμών 3 του κυρίου Μπαλτσίτη ε, να την αποσύρουμε και να στηρίξουμε την τροπολογία της κυρίας Μάρκοβατς. Ωραία. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια... Οι ερωτήσεις θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 13 ψήφοι υπέρ και μία αποχή. Εγκρίνεται η τροπολογία 6. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Ζάστε. Τέλος ψηφοφορίας. Ψήφισαν 20 υπέρ. Ομόφωνα έγινε δεκτή η τροπολογία 7. Η τροπολογία 8 έχει αποσυρθεί από το συντάκτη της. Τροπολογία 9, ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίες. 16 ψήφισαν υπέρ, 4 κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 9. Ε, μάλλον, συγγνώμη, απορρίδεται με 8 ψήφους υπέρ και 12 κατά. Τροπολογία 10 τώρα. Καταπίπτει. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. στο βοδάστ. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 4 ψήφους υπέρ και 16 κατά. Οι τροπολογίες 12, 13, 14 και 16 ψηφίζονται από κοινού. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις φυσικά να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Άρχεται η ψηφοφορία για τις τροπολογίες αυτές. Τέλος ψηφοφορίας. Γίνονται δεκτές με 19 ψήφους υπέρ και μία κατά. Τροπολογία 17. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 11 ψηφί υπέρ, 9 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 19 υπέρ, μία αποχή, εγκρίνεται. Τροπολογία 19, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Τέσσερις ψηφί υπέρ, 15 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 4 υπέρ, 16 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 17 ψήφισαν υπέρ και 2 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. 20 ψήφισαν υπέρ, παν ψηφί γίνεται δεκτή τροπολογία 2. Τροπολογία 4. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 3 υπέρ, 16 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. 13 υπέρ, 8 κατά. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για την έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Χατζημαρκάκη. Ε, Πολύ ωραία. Ο κύριος Μπαρτζίτης ψήφισε και αυτός. Και... Α, με συγχωρείτε. Ψηφίσατε ναι ή όχι κύριε Μπαρτζίτη. Έχουμε λοιπόν 20 υπέρ, 2 κατά. Έτσι και εγκρίνεται λοιπόν. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε με την ψηφοφορία για αυτή την έκθεση, τη συνάδελφοι. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Περνάμε τώρα στη συζήτηση του επόμενου θέματος στην ημερήσια διάταξη που είναι η ειδική έκθεση του ελεγκτικού συναντρίου με θέμα μπορούμε να πούμε ότι η μεταβίβαση της διαχείρισης εξωτερικής βοήθειας από τα κεντρικά γραφεία της Επιτροπής Αντιπροσωπείες οδήγησε σε βελτίωση της παροχής βοηθείας. 1 κάθετος 2011 πρόκειται και πάλι για ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Θα συζητήσουμε λοιπόν το σχέδιο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κάρελ Πίνξτεν. Α, μάλλον με διορθώνουν. Ο εισηγητής είναι ο πρώτος που πρέπει να μιλήσει. Ο κύριος Ιβάιλο Κάρτιν. Αυτός θα εισαγάγει την έκθεσή του και στη συνέχεια ο κύριος Κάρελ Πίνξτεν θα πάρει το λόγο. Λοιπόν, ο κύριος Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια έκθεση που έχει να κάνει με την απόφαση που ελήφθη το 2000 ουσιαστικά και αφορά τη χώρες περισσότερων εξουσιών στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής στα κράτη-μέλη σε σχέση με την λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή προϋπολογισμού και κονδυλίων σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτή η αποκέντρωση ξεκίνησε το 2002, το 2004 και το ελεκτικό συνέδριο πολύ σοφά αποφάσισε να ελέγξει τη λειτουργία του συστήματος μετά τη δημιουργία του και αρκετά χρόνια που πέρασαν. Εν τω μεταξύ πρέπει να σας πω ότι υπήρξε μια μεταβολή στις αντιπροσωπίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες χώρες. Δηλαδή μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατράπηκαν σε αντιπροσωπεία. Επίσης, υπήρξε μια τροποποίηση της δομής εδώ στις Βρυξέλλες με την δημιουργία της εξωτερικής υπηρεσίας και έχουμε την DG Ανάπτυξη και την EuroPaid που συγχωνεύτηκαν και φτιάξανε τη DG ETCO. Αυτές είναι όλες οι μεταβολές που έγιναν μετά το ξεκίνημα της εφαρμογής του συστήματος αποκέντρωσης. Η έκθεση συντάχθηκε για το 2009-2010 και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον το συντάκτη κύριο Πίξτον για τη, σε βάθος ανάλυση όλων των μεθοδεύσεων των αντιπροσωπιών του τρόπου λειτουργίας τους. Η έκθεση είναι πολύ συγκεκριμένη, σαφής και με σαφείς συστάσεις. Γενικά, ο κύριος Πίξτεν θα σας δώσει βέβαια τις λεπτομέρειες, αλλά γενικά λέει η έκθεση ότι η αποκέντρωση έδωσε θετικά αποτελέσματα. Βελτίωσε την ταχύτητα και την ποιότητα. Βελτίωτε, βελτίωσε την οικονομική διαχείριση και τις σχετικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα υπάρχει χώρος ακόμη για βελτιώσεις αυτών των παραμέτρων ιδίως σε σχέση με την ποιότητα της βοήθειας, την οικονομική διαχείριση, την διεύθυνση του προσωπικού στις αντιπροσωπείες και αυτές είναι συστάσεις που σίγουρα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να προχωρήσουμε με την αποκέντρωση και για να πετύχουμε μια καλύτερη υλοποίηση του προϋπολογισμού. Η έκθεση επικεντρώθηκε σε τρία ε, τρεις παραμέτρους. Την ταχύτητα χορήγησης βοηθείας, την βελτίωση της ποιότητας της βοηθείας, βοήθειας και τις διαδικασίες δημοσιονομική ε, δημοσιονομικής ε, διαχείρισης. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι η έκθεση αποτελεί θαυμάσια βάση για την Επιτροπή μας για να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση Ε, της χρήσης των πόρων για βοήθεια. Η Κομισιόν βέβαια είναι αυτή η οποία πρέπει να το φροντίσει αυτό. Σημειώνουμε λοιπόν την πρόοδο η οποία έχει ε, πραγματοποιηθεί και η Κομισιόν πρέπει να βελτιώσει τις μεθόδους αξιολόγησης ε, ώστε να αποφεύγονται μη αποδοτικά σχέδια. Και αυτό είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Δηλαδή πρέπει να αξιολογηθεί όχι μόνο η δημοσιονομική χρήση αλλά και τα αποτελέσματα της βοήθειας από τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται από τον προϋπολογισμό. Ε, υπάρχει πρακτική ε, μίσθωσης υπηρεσιών τοπικών συμβούλων και ίσως αυτή η πρακτική πρέπει να προωθηθεί για να υπάρξει παρακολούθηση της υλοποίησης των σχεδίων, της εξέλιξή τους και των αποτελεσμάτων. Δηλαδή όχι μόνο τα δημοσιονομικά αλλά και τα πρακτικά των σχεδίων πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να έχουμε αυτά ε, αποτελέσματα. Ακόμη αναφέρεται εδώ ότι η Κομισιόν πρέπει να λάβει μέτρα για να αποφύγει τα κενά τα οποία υφίστανται, ιδιαίτερα όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο. Δηλαδή ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να οργανωθεί καλύτερα όπως αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Πρέπει να δοθούν συγκεκριμένοι προσανατολισμοί στις αντιπροσωπείες από την Κομισιόν. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το προσωπικό, την επάντρωση. Αλλάζει το προσωπικό πάρα πολύ συχνά στην Γενική Διεύθυνση Συνεργασίας και Ανάπτυξης και ταυτόχρονα σε αντιπροσωπείες δεν υπάρχει προσωπικό εξειδικευμένο. Η Κομισιόν στην απάντησή της λέει ότι δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη γι' αυτό διότι η εξωτερική υπηρεσία είναι αυτή η οποία διορίζει τα άτομα, τα περισσότερα άτομα το προσωπικό δηλαδή σε αντιπροσωπεία. Όμως θα πρέπει να συνεργαστεί η Κομισιόν με την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να πετύχει αποτελέσματα. Δηλαδή θα πρέπει επιτόπου να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν πώς να οργανώσουν και να προχωρήσουν στην υλοποίηση σχεδίων. Αναφέρθηκα λοιπόν στο εσωτερικό σύστημα αναφοράς. Είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή έτσι είναι απαραίτητο να αναφέρονται τα αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνονται και υπάρχει μια πρακτική που συστήνεται στις αντιπροσωπείες για τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Όταν συζητούσαμε λοιπόν το, τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μιλήσαμε για τοπικές διαβουλεύσεις για την υλοποίηση σχεδίων σε συγκεκριμένες χώρες μαζί με τους ενδιαφερόμενους. Τέλος, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε συνέργεια η Κομισιόν να αναζητήσει καλύτερη συνεργασία με την εξωτερική υπηρεσία και με τα κράτη-μέλη. Ειδικότερα δε με, τα κράτη, ε, με τις πρεσβείες των κρατών μελών στις διάφορες χώρες ώστε να οργανωθεί η αναπτυξιακή βοήθεια μέσω των διαφορών φορέων των κρατών μελών και χρειάζεται να υπάρχει και καλύτερος συντονισμός με το έργο της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας. Ε, θυμόσαστε ότι αυτό το θέμα το συζητάμε στο Κοινοβούλιο, <coughs> την εντολή προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πρέπει πράγματι να υπάρξει ένας δεσμός, αν θέλετε, μεταξύ αυτών, διότι πολλά από τα σχέδια ε, έχουν συγχρηματοδότηση. Και οπωσδήποτε έχει γίνει κάποια δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει, δεν είναι ιδανικά τα πράγματα. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτές είναι οι βασικές συστάσεις και θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω πολύ το ελεγκτικό συνέδριο και ειδικότερα τον κύριο Πίξτεν που μας παρουσίασε μια πολύ λεπτομερή και πλήρη έκθεση. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για τις απαντώσεις που έδωσε ε, στις συστάσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Κάλφιν για το έγγραφο εργασίας που καταρτήσατε και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κάρελ Πίνξταν, που είναι το αρμόδιο μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν να κάνω την εισαγωγή σε αυτή την ειδική έκθεση, θα ήθελα δύο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω αυτή την ειδική έκθεση ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου για την Αποκέντρωση. Και επίσης να πω ότι άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τον εισηγητή σας και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω αλλά και να τον συγχαρώ γιατί διάβασα προσεκτικά την έκθεσή του και τη βρίσκω άψογη. Συγχαρητήρια λοιπόν κύριε Κάλφιν για την ε, προετοιμασία του εγγράφου εργασία σας. Οι ευρωβουλευτές μερικές φορές ε, θέλουν να μας τρομάξουν κάπως το ελεκτικό συνέδριο. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια εισαγωγή αυτή τη ειδική έκθεση, αποφεύγοντα τι επαναλήψει σε σχέση με αυτά που ήδη ακούσαμε από τον εισηγητή σα, τον κύριο Κάλφιν, σε ό,τι αφορά την αποκέντρωση. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας δώσω λίγο το ιστορικό αυτής της πρωτοβουλίας να σας πω δύο λόγια τα πορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου και να ολοκληρώσω με κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Και προχωράω στα αγγλικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το ιστορικό, το οποίο ανέφερε και ο εισηγητής σας. Ξέρετε ότι η αποκέντρωση έλαβε χώρα μεταξύ του 2002 και του 2004 και αυτή είναι η δεύτερη ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για την αποκέντρωση. Η πρώτη αυτή ειδική έκθεση ανάγεται στο 2004 ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία αποκέντρωσης και αυτή η δεύτερη ειδική έκθεση ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μία, έναν έλεγχο για την αποκέντρωση μία πενταετία και πάνω μετά την ολοκλήρωσή της. Γιατί λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο διενήργησε έλεγχο της αποκέντρωσης για τρεις διαφορετικούς λόγους. Καταρχήν, λάβαμε υπόψη την περίοδο που έλαβε χώρα, το διάστημα που μεσολάβησε από την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων στις αντιπροσωπείες. Δεύτερον, Επειδή τότε κρεμούσε ακόμη η θέσπιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που στο μεταξύ έχει τεθεί σε εφαρμογή και επίσης γιατί 80% της ε, βοήθειας που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, περνάει μέσα από το αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης πια. 80% αυτής της ε, ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περνά μέσα από τις αντιπροσωπείες τελικά ως προς τη διαχείριση. Η ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο της αποκέντρωσης ασχολήθηκε με την ταχύτητα, της, ε, την ποιότητα της χορήγησης ενίσχυσης αλλά και τη δημοσιονομική ε, διαχείριση. Κατά πόσο οι διαδικασίες αυτής της δημοσιονομικής διαχείρισης ήταν ε, δρεωμένες και στεναρές και ή όχι. Σε αφορά την ταχύτητα, το πρώτο σημείο, την ταχύτητα χορήγηση τη ενίσχυση. Όπως είπε και ο εισηγητή σα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να δεσμεύσει και να καταβάλει πολύ μεγαλύτερα ποσά ενίσχυση ε, μετά την εφαρμογή της αποκέντρωσης. Και αυτό το θέμα ε, απασχόλησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί προβλήματα που είχαμε πριν την αποκέντρωση με συσσόρευση ποσών το έχουμε ξεπεράσει με την αποκέντρωση. Βέβαια η ταχύτητα μπορεί να βελτιωθεί και περαιτέρω, ταχύτητα της χορήγησης, με πιο συγκεκριμένες ε, προτάσεις και συστάσεις. Πάντως θεωρούμε ότι η ταχύτητα της χορήγησης της βοήθειας ε, έχει βελτιωθεί αισθητά. Αυτά ως προς τη ταχύτητα. Τώρα σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές διαδικασίες. Θεωρούμε ότι και εδώ Υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις των διαδικασιών δημοσιονομικής διαχείρισης και μάλιστα προφανείς βελτιώσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τρίτο σημείο, την ποιότητα της ε, παρεχόμενης ενίσχυσης, αυτό το θέμα της ποιότητας της βοήθειας δεν είναι και τόσο προφανές. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η ποιότητα της βοήθειας έχει βελτιωθεί. Ναι μεν, αλλά διαπιστώνουμε ότι το σύστημα καταμέτρησης αυτής της ποιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μας δίνει μια περιεκτική εικόνα, μια συνολική εικόνα που μας επιτρέπει να ε, συναγάγουμε κάποια αδιάσυστα συμπεράσματα. Αυτή τη στιγμή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο εξωτερικό σύστημα ROM, που είναι το σύστημα αξιολόγησης προσανατολισμένο στα αποτελέσματα, παρακολούθηση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Θέλουμε μια πιο τεκμηριωμένη και διεξοδική αξιολόγηση της ποιότητας της βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό προβαίνουμε σε δύο συστάσεις στην ειδική μας έκθεση. Καταρχήν, πιστεύουμε ότι οι αντιπροσωπείς θα πρέπει να διεξαγάγουν και αξιολογήσεις της αποδοτικότητας όλων των παρεμβάσεων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν και ποσοτικές ε, εκτιμήσεις. Όχι μόνο ποιοτικές αξιολογήσεις, αλλά και ποσοτικές καταμετρήσιμες αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων αυτού, αυτής της ε, βοήθειας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διαδικασίες δημοσιονομικής διαχείρισης. Ο έλεγχος μας επισήμανε τρεις τομείς, στους οποίους επιστούμε και την προσοχή της Επιτροπής. Καταρχήν, ε, το θέμα της αναφοράς ε, της ε, έκθεσης και του ελέγχου στα θέματα διαχείρισης, το ρόλο των ε, αρχηγείων κατά κάποιο τρόπο, των κεντρικών γραφείων συνεργασία και το θέμα της πρόκλησης που δημιουργεί η συνεχής εναλλαγή των ανθρωπίνων πόρων. Στην δική μας έκθεση υποβάλλουμε κάποιες συστάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των τριών τομέων σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση, την ενημέρωση και την αξιολόγηση. Η παρακολούθηση σε επίπεδο αντιπροσωπείας θα πρέπει να γίνεται συστηματικά σε μια γενική στρατηγική παρακολούθηση για κάθε αντιπροσωπεία. Επίσης πιστεύουμε ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και ενημέρωσης θα πρέπει να ε, είναι προσανατολισμένο περισσότερο στα αποτελέσματα των διαφόρων παρεμβάσεων και σε ό,τι αφορά την, την ίδρυση τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, οι νέε διατάξεις για τη λογοδοσία των επικεφαλή των αντιπροσωπιών θα πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Τώρα, ο ε, ε, ενισχυτικό και βοηθητικός ρόλος των κεντρικών γραφείων. Όπως είπε ο κύριο Κάλφιν, ο μεγάλος βαθμός ε, εναλλαγής του προσωπικού στο Γραφείο Συνεργασίας της EuroPaid θα πρέπει να ληφθεί υπόψη γιατί δημιουργεί προβλήματα και χρειάζομαστε και περισσότερες ε, οδηγίες ό,τι αφορά το διάλογο για τις πολιτικές. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί ο διάλογος για τις πολιτικές είναι πολύ σημαντικό θέμα στα πλαίσια της δημοσιονομικής διαχείρισης. Και τώρα σε ό,τι αφορά την πρόκληση για τους ανθρωπίνους πόρους. Είναι σημαντικό να έχουμε την αξιοποίηση, την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προσωπικού με στόχο την μηδενική αύξηση του προσωπικού. Αυτό το λάβαμε υπόψη και το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να μην διευρύνει το προσωπικό της μέχρι το 2013, για μια εξαιτία δηλαδή, να μην προσλάβει νέους υπαλλήλους και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνει καλύτερη κατανομή του υφιστάμενου προσωπικού. Και αυτό το θέμα τη σωστή ιδεώδου κατανομής και τη αξιοποίηση είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πενιχρή η ανθρώπινη πόλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, λιγομελές στο προσωπικό και θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως αναφέρεται και στην ειδική έκθεση. Δύο είναι οι συστάσει μα σχετικά. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει την παρούσα χρήση του το προσωπικού ώστε να εξασφαλίσει ε, τη σωστή χρησιμοποίηση του και αξιοποίηση του προσωπικού και να υπάρχει προσωπικό και πραγματικά χρειάζεται γιατί πραγματικά είναι ελάχιστο το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συνιστούμε να έχει στενότερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να μειωθούν οι τομεί παρέμβαση στι οποίε συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ζητούμε επίση να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία των κρατών μελών. Και έρχομαι τώρα στις ε, καταληκτικές μου παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω, όπως είπα, τον εισηγητή σας για τα σχόλια που υπέβαλε και τα δέχομαι εκ μέρους και της ομάδας μου, το επιτελείο μου που κατήρτισε την ειδική αυτή έκθεση για την αποκέντρωση και φυσικά δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου χωρίς να επενέσω τη θετική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή την θετική στάση. Φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Όσον αφορά τις ε, ειδικέ εκθέσεις, ε, θα ήθελα να ανοίξουμε τη συζήτηση και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κρέσλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω και εγώ τις δικές μου ευχαριστίες γιατί αυτή είναι μια πολύ σημαντική έκθεση και είναι από τις, μια από τις ελάχιστες διαθέσιμες εκθέσεις που ασχολούνται με το θέμα της αποκέντρωσης μετά τη μεταρρύθμιση στην οποία προέβη η Κομισιόν. Και νομίζω ότι είναι και η μοναδική έκθεση που αφορά το πώς ακριβώς ε, επέδρασε το θέμα της ε, αποκέντρωσης. Και επειδή είναι λοιπόν η μόνη διαθέσιμη έκθεση, πρέπει να πω, λυπάμαι πάρα πολύ που η έκθεση δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία. Η έκθεση αυτή δεν λέει τίποτα για τα θέματα της ενίσχυσης. Ε, κυρίως ε, δεν αναφέρεται στο τι συνέβη κατά το παρελθόν. Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε κάτι τέτοιο. Αυτό δηλαδή που θέλω να πω είναι το εξής. Η μετάταξη προσωπικού από ε, τις περιφερειακές, τις περιφερειακές οργανώσεις στο κεντρικά, στα κεντρικά γραφεία αυτό δεν ε, παρουσιάζεται καθόλου. Ε, στην γερμανική τουλάχιστον μετάφραση, στη σελίδα 10, στο γράφημα υπαριθμών 1, αν δει κανεί τις μετακινήσεις από τις αντιπροσωπείες στα κεντρικά γραφεία, καταλήγει κανείς το συμπέρασμα ότι τελικά όλη αυτή η διαδικασία χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία και δισκαμψία. Αυτό λοιπόν προκύπτει από αυτό το γράφημα και θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια το ελεγκτικό συνέδριο για αυτό το γράφημα γιατί νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό και να το αναλύσουμε ενδελεχώς. Τώρα, όσον αφορά την ΤΕΦΚΟ, η ΤΕΦΚΟ εξακολουθεί να έχει 2.500 ε, υπαλλήλους. Και αυτό το βρίσκω πολύ ιδιαίτερα εντυπωσιακό τον αριθμό. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να μάθουμε τι ακριβώς προέβη, τι προέκυψε με την ε, μετάταξη των υπαλλήλων. Αυτό είναι το πρώτο που επιθυμώ. Το δεύτερον, αν δει της αντιπροσωπής τις 163 που έχουμε εντωμεταξύ και εκεί βλέπω ότι υπάρχει κάποια αυθαιρεσία στην κατανομή προσωπικού. Η κατανομή προσωπικού δεν προσαρμόζεται στο ποσό. Δηλαδή έχουμε αντιπροσωπείες που έχουν 60 ανθρώπους και δαπανούν 5 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε αντιπροσωπείες που έχουν και αυτές 60 άτομα αλλά δαπανούν το 1 τρίτον των 60.000 και οι δύο ασχολούνται με δύσκολα θέματα. Άρα δηλαδή που δεν είναι δικαιολογείται στη μία αυτή η υπερβολική αύξηση του ποσού. Και ακούω βέβαια ότι εντωμεταξύ ε, καμία αντιπροσωπεία ή ε, κανένας οργανισμός δεν θέλει να του αφαιρέσουν προσωπικού γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι θέμα γοήτρου. Είναι δηλαδή γόητρο το να έχει πολλούς υπαλλήλους. Ε, πρέπει να τα εξετάσουμε λιγάκι όλα αυτά και θα ήταν σημαντικό το ελεγκτικό συνέδριο να μας προσφέρει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Κατόπιν το θέμα του προϋπολογισμού κυρίως budget support όπως αναφέρεται. Ε, εδώ αναφέρεται λεπτομερώς το ελεγκτικό συνέδριο στο θέμα αυτό και του είμαι ευγνώμων. Ε, θεωρώ ότι και αυτό, όπως και το θέμα του προσωπικού, πρέπει να το επανεξετάσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε ε, να εκταμιεύει όλο και περισσότερα χρήματα. Ε, αυτή τη στιγμή ε, δαπανά το ίμιση αυτό που θα έπρεπε, εκταμιεύει το ίμιση αυτό που θα έπρεπε, όμως η τάση είναι αυξητική. Και τίθεται το εξής ερώτημα. Τι θα γίνει στο μέλλον. Εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε να επεκτείνουμε το budget support, αλλά η Κομισιόν σε εθνικό επίπεδο αποφασίζει κάτι άλλο. Και ρωτώ την Κομισιόν πώς μπορεί κανείς να τα συνδέσει αυτά τα δύο ε, μήπως ε, σημαίνει όλο αυτό ότι δεν λαμβανόμεθα σοβαρά υπόψη σε αυτά που αποφασίζουμε. Στην επόμενη επαλλαγή θα πρέπει να επανέλθουμε τι θα γίνει με το budget support και τι προβλέπετε για την εκπαίδευση των υπαλλήλων έτσι ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε την στήριξη του προβλογισμού, το budget support, όπως ακριβώς προβλέπετε. Κάτι άλλο που ε, θα έπρεπε να εξετάσουμε είναι τι θα γίνει ε, με την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η οποία έχει πολύ λιγότερους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ περισσότερα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε αν τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να προσλάβει και άλλο προσωπικό. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς αυτό σημαίνει. Αυτή είναι μια ε, πολύ σημαντική έκθεση και εκείνο που δεν βλέπω είναι να υπάρχει μια ποσοτικοποίηση Δηλαδή, ε, πώς ακριβώς βελτιώθηκε η βοήθεια που παρέχουμε. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες ε, του ελεγκτικού συνεδρίου ε, όλα αυτά να εκφραστούν ποσοτικά με αριθμούς. Ας πούμε, ε, μέχρι τώρα τίθεται το ερώτημα πόσα ανεπαρκή προγράμματα υπήρξαν. Το 2004 4%, το 2009 6%. Είναι 6%, είναι σημαντικό το ποσοστό αυτό. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα μπορούμε να μειώσουμε το ποσοστό αυτό. Τι είδους άλλους δείκτες έχουμε. Στο γράφημα υπερθμών 5 βλέπουμε ότι μειώνεται το θέμα της αηφορίας και στην αποτελεσματικότητα και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια αύξηση, έστω και μικρή αύξηση όμως είναι αυτή. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει η βέλτιστη χρήση των κονδυλίων και μήπως πρέπει να προσπαθήσουμε να ποσοτικοποιήσουμε περισσότερο τη βοήθεια. Είμαι λιγάκι κριτική σε όλα αυτά γιατί ο τομέας αυτός που ε, βρίσκεται μπροστά σε μια τεράστια αναδιάρθρωση, τον τομέα αυτό θα πρέπει να τον εξετάσουμε προσεκτικότερα κατά τα επόμενα έτη και μπορούμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε το ελεγκτικό συνέδριο ε, το νέο αυτό οικοδόμημα να το αντιμετωπίσει με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως και το παλαιό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας. Ε, μήπως υπάρχει κάποιος ε, ο οποίος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Αν όχι, θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν υπάρχει κάποιος που επιθυμεί να λάβει το λόγο και θέλει να συμβάλλει στη συζήτηση. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεση του. Θαυμάσια έκθεση και ευχαριστώ για την έκθεση αυτήν τον κύριο Καλφίν. Ε, κάναμε και τις δικές μας αναλύσεις πρέπει να σας πω. Είναι πολύ επίκαιρη λοιπόν αυτή η έκθεση επειδή ο Επίτροπος μας θέλει να ανασχεδιάσουμε την αναπτυξιακή πολιτική. Επίσης στην αρχή του έτους δημιουργήθηκε η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχουμε και την ε, Διεύθυνση Πολιτικής και υπάρχει και κάτι καινούργιο που ίσως δεν σημειώσαμε. Η νέα Γενική Διεύθυνση αναλαμβάνει κάποιες εξουσίες σε σχέση με το προσωπικό που, βρίσκονται στη, που βρίσκεται στις αντιπροσωπείες. Είναι η πρώτη φορά που η Γενική Διεύθυνση λοιπόν στην έδρα έχει την ευθύνη και για το προσωπικό επιτόπου συμφωνούμε με τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου συνολικά καθώς και με τις συστάσεις του εισηγητή κύριε Μπάλκη. Ε, επιτρέψτε μου κάποια σχόλια. Όσον αφορά την οικονομική διαχείριση, από το 2002 συνεχώς βελτιώσαμε τα συστήματα ελέγχου και εποπτείας. Το ελεγκτικό συνέδριο άλλωστε αναφέρει στην έκθεση ότι έχουμε ένα ποσοστό λαθών μη ανευσημασίας, πράγμα το οποίο καταδεικνύει την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά την ποιότητα επίσης από το 2002, εκ παραλλήλου με την εφαρμογή της αποκέντρωσης, έχουμε εισαγαεί και συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας. Αυτό ευεξηγεί τον προς πίσω που υπάρχει, αν θέλετε, μεταξύ αντιπροσωπείας και έδρας η έδρα υποστηρίζει τις αντιπροσωπείες στην ταυτοποίηση των σχεδίων και γι' αυτό πηγαίνω έρχονται αν θέλετε τόσο έγγραφα, τόσο έγγραφα μεταξύ έδρας και αντιπροσωπείας. Ε, το επίπεδο της ποιότητας δεν μπορούμε να το μετρήσουμε πολύ απλά. Έχουμε βεβαίως το Result Monitoring System. Ε, μετράμε βασικά όμως τα αποτελέσματα. Και αν θέλετε αυτό είναι μια η μέτρηση δηλαδή των αποτελεσμάτων είναι μια πρόκληση, εξακολουθεί να είναι πρόκληση. Όσον αφορά την διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, σας είπα προηγουμένως ότι έχουμε μια νέα γενική διεύθυνση, την ΤΕΦΚΟ, που έχει την άμεση ευθύνη του προσωπικού που βρίσκεται σε αντιπροσωπείες. Θα έπρεπε λοιπόν αυτή η Γενική Διεύθυνση να μπορέσει να εξομοιώσει, να ισορροπήσει μάλλον καλύτερα τις ανάγκες και τους πόρους, ε, λαμβάνοντα υπόψη τη μηδενική αύξηση των ανθρωπίνων πόρων στην Κομισιόν. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία αξιολόγηση του έργου των αντιπροσωπιών. Ακολουθούμε μία ενδεδειγμένη μεθοδολογία και θα έχουμε τα αποτελέσματα περίπου τον Νοέμβριο. Αυτή η αξιολόγηση θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε ένα πολυετές πρόγραμμα ώστε να έχουμε σωστή ανάπτυξη του δυναμικού μας από την άποψη του προσωπικού. Επίσης η συνεργασία με τους φορείς των κρατών μελών είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά για να χορέψει κανείς το τάγκο πρέπει να, είναι, να είμαστε δύο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κατανομή της εργασίας μόνοι μας. Χρειαζόμαστε να έχουμε συμμετοχή. Έχουμε βελτιωθεί από το 2002, έχουμε υιοθετήσει με τα κράτη-μέλη λοιπόν, ένα κώδικα για την κατανομή του, των εργασιών, αλλά χρειαζόμαστε πρόσθετες προσπάθειες ώστε η κατανομή και του έργου και των εργασιών ε, να είναι πιο αποτελεσματική στο επίπεδο της Ένωσης πλέον. Όσον αφορά τώρα τις χορηγίες και τα δάνεια, και την αποκοινού χρησιμοποίησή τους. Η Κομισιόν συμφωνεί με την προσέγγιση, άλλωστε έχει δεσμευτεί εδώ και μερικά χρόνια με τη δημιουργία του Ταμείου Ανάπτυξης για τις χώρες ΑΚΕ και με τη δημιουργία του Μηχανισμού Γειτονίας Λοιπόν, αυτά είναι, αν θέλετε, μηχανισμοί που θέλουμε να αναπτύξουμε, αν συμφωνήσει η αρχή για τον προϋπολογισμό. Ε, Βεβαίω όμως αυτοί οι μηχανισμοί πρέπει να υπάγονται στην πολιτική για την ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και πάλι το ελεκτικό συνέδριο για το έργο του. Συμφωνούμε με την ανάλυση που έχει κάνει και θα εφαρμόσουμε τις συστάσεις που εγκρίνατε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν, για τη συμμετοχή στη συζήτηση. Κυρία Γκρέσλε. Η Κομισιόν αλλά ούτε και το ελεγκτικό συνέδριο απάντησαν στην ερώτηση που έτσι Απλά ήθελα να το επισημάνω αυτό. θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πίνξτεν ε, για να απαντήσει αν μπορεί. Κύριε Πίνξτεν, μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε. Και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάλφιν, τον εισηγητή μας, για να ανακεφαλώσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος με τις παρατηρήσεις που έκανε η κυρία Γκρέσλε γιατί πραγματικά η κυρία Γκρέσλε επισήμανε, έθεσε το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων, επισήμανε τα πραγματικά προβλήματα που έχουμε. Θα βρείτε και τα αποτελέσματα του ελέγχου στην ειδική έκθεση και τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδριού. Εννοείται όμως ότι και το ελεκτικό συνέδριο θα δώσει μια συνέχεια στις συστάσεις, θα παρακολουθήσει την ε, εφαρμογή των συστάσεων. Χαίρομαι μεν που η ειδική έκθεση έτυχε τέτοια ενθουσιώδους υποδοχής και από το Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα συνεχίσουμε την παρακολούθηση για να δούμε αν όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη και εφάρμοσε τις συστάσεις μας. Και συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Γκρέσλε, δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που είπε, γιατί σε επίπεδο προσωπικού υπάρχουν κενά, θα πρέπει να γίνουν πολλές προσπάθειες και ακόμη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη εκεί. Το ελεκτικό συνέδριο βέβαια δεν είναι πολιτικό όργανο όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή κάπως πολιτικό όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξαρτάται και από το χαρτοφυλάκιο του κάθε επιτρόπου. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπα και στην εισαγωγή μου προηγουμένως για την παρουσίαση της ειδική έκθεσης, είναι ευνόητο ο Ευρωπαίος φορολογούμενος να απαιτεί ε, ο αρμόδιος επίτροπος να έχει συζήτηση και διάλογο με τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την κατανομή και τον καταμερισμό του έργου. Γιατί άλλες χώρες έχουν περισσότερο προσωπικό ή άλλες υπηρεσίες και άλλες λιγότερο. Καλό είναι να υπάρχει ένα συντονισμός και μια συνεργασία. Και ούτε όλες οι αντιπροσωπείες έχουν το ίδιο προσωπικό, τον ίδιο αριθμό των υπαλλήλων. Και εκεί θα πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Ο πίνακα 1 που μιλάει για το καταμερισμό των ευθυνών είναι φω φανάρι και επαναλαμβάνει το αίτημα τη κυρία Γκρέσλε. Έχουμε μια ολόκληρη σελίδα. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω καν τον όρο γραφειοκρατία, δεν είμαι εγώ αρμόδιο να το κάνω, αλλά βλέπετε μια ολόκληρη σελίδα με αυτά που επισημάνατε και εσείς κυρία Γκρέσλε. Σε ό,τι αφορά τώρα την ποσοτικοποίηση της ποιότητας, την καταμέτρηση της ποιότητας με αριθμούς. Και ω προ την διαδικασία δημοσιονομική διαχείριση, νομίζω ότι είναι απερίφραστα τα συμπεράσματα. Σε ό,τι αφορά την επιτάχυση τη βοήθεια. Και εκεί τα συμπεράσματα είναι ξεκάθαρα. Αλλά όπω είπα και στην εισαγωγή μου, στα θέματα ποιότητα τη βοήθεια, εκεί στο μέλλον υπάρχει δυνατότητα καταμέτρησης, ποσοτικοποίησης των αποτελεσμάτων και αποτίμηση της ποιότητας της βοήθειας. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ίσως το ξέρουν αυτό εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εμείς το γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο βοήθειας ε, στις περισσότερες χώρες του κόσμου είναι ο υπαριθμόν ένα χορηγός ενίσχυσης. Δεν είναι ψυχία αυτά που δίνουμε. Είμαστε ο, ο πρωταρχικός δωρητής βοήθεια στον τρίτο κόσμο, ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλου είδους αρρωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπαριθμών ένα χορηγός και λογικό είναι να κάνουμε όσες προσπάθειες γίνεται, να ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις καταβάλει. Και όπως είπε και η κυρία Γκρέσλε, φυσικά υπάρχει δυνατότητα ποσοτικοποίησης, ε, καταμέτρησης της ποιότητας. Για να διαπιστώσουμε αν όντως υπάρχει βελτίωση, αναβάθμιση της ποιότητας είναι πολύ πιο εύκολο να αποτιμήσουμε την ποιότητα εφόσον μπορούμε να την ποσοτικοποιήσουμε. Και εκεί όντω πρέπει να γίνει μια περαιτέρω προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστώ πάντω γιατί ήταν πολύ εύστοχα τα σχόλια, πολύ τεκμηριωμένα και ευγενικά όπω συνήθω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Κόφιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι εγώ δεν έχω να προσθέσω πολλά. Ήταν θαυμάσια η έκθεση. Παρουσίασε με απόλυτη σαφήνεια τις ε, συστάσεις. Έχουμε θετική αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα δηλαδή αυτές θα ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στο τέλος ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε ότι επιθυμεί να βελτιώσει την ποιότητα και όλη αυτή τη διαδικασία παροχής αναπτυξιακής βοήθειας. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς. Μιλάμε για θέματα τα οποία ε, είναι εκτενή και πολλές φορές όμως εμείς ε, δημιουργούμε προηγούμενο. Οι απαντήσει δεν είναι πάντα σαφείς. Όταν μιλάμε δηλαδή για την ποιότητα της αναπτυξιακής ε, βοήθειας, αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να μας ενδιαφέρει, η ποιότητα. Και βεβαίως ε, στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και ο κύριο Πίνξτερ το είπε με απόλυτη σαφήνεια, είναι σαφέ ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη καταμέτρηση και αποτίμηση της ε, ποιότητας. Οποτεδήποτε μιλάμε για αναπτυξιακή βοήθεια, δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε όλα με αριθμούς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες. Αλλά δεν πρέπει και να περιμένουμε ότι ε, θα έχουμε μία αριθμητική απεικόνηση μπροστά μας ως εξήγηση. Ε, θα ήμουν λοιπόν ιδιαίτερα ευτυχής ε, αν η Κομισιόν ε, παρουσιάζοντας τα ποιοτικά κριτήρια μπορούσε στο Κοινοβούλιο να μας ε, παρουσιάσει και την ευρύτερη ε, νοοτροπία και το πώς προβλέπεται να ο έλεγχος στην ποιότητα. Υπάρχει θέμα συντονισμού ανάμεσα στους διάφορους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ανάμεσα στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή. Γνωρίζουμε ότι αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί μακράν αυτού και εξακολουθούμε να κάνουμε τα βήματα εκείνα τα οποία εν ευθέτω χρόνο θα οδηγήσουν σε καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στους ε, δύο θεσμούς. Μιλάμε επίσης ε, και συντονισμό με τους εξωτερικούς δωρητές. Ε, σωστό αυτό. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια ε, προφανώς έρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα κράτη-μέλη, αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι δωρητές, αλλά θα πρέπει και πάλι να έχουμε κατά νου ότι αυτή η διαδικασία, γιατί βέβαια συζητάμε για διαφορετικά θέματα, ε, αυτά έχουν σχέση με την διαφάνεια, ε, το κατά πόσο είναι ορατή η αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτά δεν είναι εύκολο να τα λύσει κανείς οποτεδήποτε συνεργάζεται με άλλους θεσμούς. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι πολύ σωστά πράξαμε να επεκτείνουμε την αναπτυξιακή βοήθεια. Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά που είπε η κυρία Γκρέσλε και τα σχόλιά της και τα στηρίζω, διότι η αύξηση των ε, εκταμιευόμενων κονδυλίων, αυτή η αύξηση είναι συνάρτηση και του αυξημένου ελέγχου. Είδατε, στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αναφέρεται σαφής μείωση των μη αποδοτικών προγραμμάτων που σημαίνει ότι ακόμα και όταν εκμεταμιεύονται τα απαραίτητα κονδύλια πρέπει να υπάρχει μια σωστή εξέλιξη. Το θέμα της ποιότητας λοιπόν είναι καθοριστικής ε, σημασίας ε, και οι προεκτάσεις της αναπτυξιακής βοήθειας. Θέλω όμως να σας προειδοποιήσω να μην υπάρχουν ε, υπερβολικές ε, προσδοκίες και να μην θέλουμε όλα να εκφράζονται αριθμητικά. Εγώ στηρίζω αυτά που είπε ο κ. Πίνξτεν ότι πράγματι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το παρακολουθήσουμε και στο μέλλον καθότι ε, τα προβλήματα τα οποία αγγίζει είναι προβλήματα τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τα τεχνική φύσεως θέματα που παρουσιάζονται σε άλλου είδους εκθέσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Κάλφιν. Κυρίε και κύριοι, ολοκληρώσαμε το σημείο 7 της ημερήσης διάταξης και μπορούμε το σημείο 6 συγγνώμη, της ημερήσης διάταξης και μπορούμε να περάσουμε στο τελευταίο για σήμερα θέμα, το σημείο 7 που προβλέπει την ανταλλαγή απόψεων για την ειδική έκθεση του Ενεκτικού Συνεδρίου Περθών 2 του 2011 παρακολούθηση της ειδική έκθεσης ε, παριθμών 1 του 2005 σχετικά με τη διαχείριση της ΟΛΑΦ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης. Ο υποφαινόμενος είναι ο εισηγητής για το θέμα αυτό. Και τώρα πια έχω πολλές ιδιότητες ταυτόχρονα, γιατί δεν είμαι μόνο ο πρόεδρος της Επιτροπής σήμερα, αλλά είμαι και ο εισηγητής αυτής της έκθεσης. Άρα, μια και δεν έχω άλλη επιλογή, θα δώσω εγώ το λόγο στον εαυτό μου. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα χωρίς να είμαι υπερβολικά αυρόφρον και εγκομιαστικός, ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λουί Γκαλέα και τους συνεργάτες του για την διεξοδική και πολύ τεκμηριωμένη ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και πριν περάσουμε στην ανταλλαγή απόψεων θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ τους, και τους εκπροσώπους της και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν έχετε μανία με τα νούμερα, θα, και τις στατιστικές, θα δείτε ότι η πρώτη έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου καταρτίστηκε πέντε χρόνια μετά την ίδρυση της ΟΛΑΦ. Και πέντε χρόνια αργότερα έχουμε τη δεύτερη πια έκθεση, δεύτερη ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου, που ήταν η συνέχεια της πρώτης, πρώτη 2005, η δεύτερη το 2011 και θέμα η ανάλυση για το κατά πόσο η ΟΛΑΦ έλαβε υπόψη τις συστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου. Και αν το Ελεκτικό Συνέδριο έχει αυτή την πρόθεση να ερευνά τι γίνεται στην ΟΛΑΦ κάθε πέντε χρόνια, εντάξει, αλλά νομίζω ότι είναι σύμπτωση που συνέβη αυτό κάθε πέντε χρόνια. Πάντως, είναι σημαντικό να προβαίνουμε τακτικά σε αξιολόγηση του έργου ενό πολύ σημαντικού οργάνου, όπω είναι η ΟΛΑΦ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κατά Πολέμη Απάτη. Η αρχική έκθεση του ερεκτικού Συνεδρίου περιλάμβανε 17 συστάσει που θα μπορούσαμε να τι ταξινομήσουμε σε τρει κατηγορίε. Το πιο σημαντικό θέμα ήταν η ενίσχυση των ερευνητικών λειτουργιών τη ΟΛΑΦ και το κατά πόσο μπορεί ο ΛΑΦ να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της και να αποδείξει την αποδοτικότητα των ερευνών της. Επίσης, ε, οι αδυναμίες διαχείρισης της ΟΛΑΦ που είχαν αντοπιστεί στην πρώτη ειδική έκθεση, πώς είναι δυνατόν ε, να διορθωθούν και να ξεπεραστούν. Το δικό μου έγγραφο εργασία αναγνωρίζει το μέχρι τώρα έργο της Όλαφ που επιτέλεσε από, στο διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη έκθεση μια πενταετία, δηλαδή εξαετία μετά τον εντοπισμό των προβλημάτων φαίνεται ότι η ΟΛΑΦ κατάφερε να βελτιώσει την ποιότητα του έργου της και μάλιστα ίδρυσε και δύο ε, γενικές διευθύνσεις έρευνας, ενώ είχε μόνο μία και αύξησε τον αριθμό των επιτόπιων ε, ελέγχων και ερευνών, βελτίωσε το λογισμικό της, περιόρισε τα περιθώρια σφάλματος και μείωσε και του συμβασιούχους της στο προσωρινό προσωπικό. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα διαχείρισης που ακολούθησαν τις ε, συστάσεις της πρώτης ειδική έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου για την ΟΛΑΦ. Η δεύτερη ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου διαπιστώνει ότι από τις 17 αρχικές συστάσεις της πρώτης ειδικής έκθεσης, 14 ελήφθησαν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφαρμόστηκαν στην ΟΛΑΦ και από τις 14 αυτές συστάσεις που κρίθηκαν χρήσιμες, από τις 14 αυτές λοιπόν συστάσεις που κρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρήσιμες, μόνο τρεις εφαρμόστηκαν πλήρως στο έργο της ΟΛΑΦ. Δεν ναι, μεν τις έκρινε χρήσιμες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τις εφάρμοσε. Μόνο τρία τέταρτα λοιπόν των πολύ χρήσιμων συστάσεων του ελεκτικού συνεδρίου ε, αγνοήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί μόνο ε, λίγες συστάσεις εφαρμόστηκαν. Το νέο έγγραφο είναι η ειδική έκθεση, περιλαμβάνει εννέα συστάσεις και επειδή ακριβώ μας πιέζει ο χρόνος αλλά και επειδή σας είχαμε μοιράσει εγκαίρως το έγγραφο εργασία. δεν πρόκειται να υπησέλθω σε διεξοδική ανάλυση αυτών των συστάσεων θα επικεντρωθώ σε τρεις μόνο από αυτές που κατά τη γνώμη μου είναι και οι πιο σημαντικές. Ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι η μέση διάρκεια διαλέπκες μιας υπόθεσης είναι μια διετία και αυτή η διάρκεια δεν έχει βελτιωθεί δεν έχει βελτιωθεί ο μέσος όνος διεκπαιρέωσης μια, μιας υπόθεσης. Μια χρονοτριβή που είχε επισημανθεί στην πρώτη ειδική έκθεση. Και μάλιστα μόνο το 37% των ε, ερευνών ε, είχαμε για το 2009. Θα πρέπει να βελτιωθεί αυτό το ποσοστό. Μόνο 37% ήταν η διεξαγωγή ερευνών από το συνολικό χρόνο της ε, υπηρεσίας της ΟΛΑΦ. Επίσης και η αρχική φάση της ε, διερεύνησης μιας υπόθεσης διπλασιάστηκε από 3,5 μήνες. Αυτή η αρχική φάση κρατάει πια 7 μήνες. Αυτό βέβαια οφείλεται σε μια γενική παράταση του ερευνητικού χρονικού πλαισίου για τη συγκέντρωση των πληροφοριών. Χρειάζεται πια περισσότερος χρόνος από ό,τι φαίνεται, διπλάσιος πια χρόνος. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι μέσα αυτό το επτάμινο έγινε σημαντικό διερευνητικό έργο, χωρίς όμως τις εγγυήσει που δίνει μια τακτική ερευνητική διαδικασία. Μία άλλη σύσταση της έκθεσής μου που αντιγράφει ουσιαστικά σύσταση της ειδικής έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου επισημαίνει την έλλειψη ανεξάρτητου μηχανισμού ελέγχου και επισημαίνει και κάποια διαδικαστικά προβλήματα. Είναι σημαντικό να διορθωθεί αυτή η κατάσταση από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται δηλαδή ένα νομοθετικό έργο για να ξεπεραστούν αυτές οι αδυναμίες και να θεσπιστούν κάποιες νομικές διατάξεις χωρίς όμως να μεταρρυθμιστεί ολόκληρο το νομικό πλαίσιο της ΟΛΑΦ. Γιατί μόνο με τέτοιες ε, αλλαγές ε, κάποιων νομοθετικών διατάξεων θα βελτιωθεί και η αποτελεσματικότητα των εργασιών της ΟΛΑΦ. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω λοιπόν το αρμόδιο μέρος του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Γκαλέα, για το έργο του στην κατάρτιση της ειδικής αυτής έκθεσης και να καλωσορίσω στη συνεδρίασή μας και εκπροσώπους της ΟΛΑΦ και να περάσουμε στην ανταλλαγή των απόψεων. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Γκαλέα, εκ μέρους του Ελεκτικού Συνεδρίου. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους του Ελεκτικού Συνεδρίου θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω πόσο εκτιμούμε την πρόσκλησή σας που μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις διαπιστώσεις και για την έκθεση παρακολούθησης. Η αρχική έκθεση του 2005, όπως αναφέρατε, είχε υποβάλει 17 συστάσεις που αναφερόντουσαν σε διάφορες πτυχές της λειτουργίας της Όλαφ. Με βάση λοιπόν αυτές τις συστάσεις, το δικαστήριο έκανε τον έλεγχό του και την κριτική του ανάλυση. Θα ήθελα όμως ταυτόχρονα να απογραμμίσω το γεγονός ότι η περίληψη της έκθεσης του συντάκτη της δικιάς σας ε, έκθεσης ε, είναι πάρα πολύ καλή, αναφέρεται στις διαπιστώσεις κλειδιά. Διαβάσαμε σε βάθος την έκθεσή σας και συμφωνούμε με τα σχόλιά σας, καθώς και με τη σύστασή σας να περιληφθούν αυτές οι συστάσεις στην απαλλαγή ε, της Κομισιόν για το 2010. Θα ήθελα με την ευκαιρία να υποστηρίξω το έργο των ελεγκτών του ελεκτικού συνεδρίου για τη σύνταξη αυτή της έκθεσης. Βοήθησαν πολύ. Κάναμε μια κριτική ανάλυση λοιπόν του τρόπου διοίκησης και των λειτουργιών της Όλαφ. Και θέλουμε ακόμη να αποσαφηνίσουμε ότι αυτό το πράξαμε επειδή είμαστε πεπισμένοι για τη σπουδαιότητα της Όλαφ της ίδιας είναι σημαντικό το έργο της Όλαφ, επαναλαμβάνω. Και ακριβώς εκτιμούμε ιδιαίτερα και το φόρτο εργασίας, αλλά και το δύσκολο έργο που, έχουν πολύ που παράγουν πολλοί ελεγκτές της Όλαφ, και αν θέλετε δεν θέλω, ε, να μακρηγορήσω, η συγκητής ήδη μας υπενθύμησε την εφαρμογή των συστάσεων του 2005, τον τρόπο που εξελίχθησαν κτλ. Οι περισσότερες από αυτές τις συστάσεις λοιπόν εφαρμόστηκαν σε διαφορετικό βαθμό και γι' αυτό το δικαστήριο θα ήθελε να επαναλάβει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες συστάσεις του. Συνεπώς πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των συστάσεων. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε τρία σημαντικά μηνύματα που προκύπτουν από τις διαπιστώσεις του δικαστηρίου. Πρώτον, η Όλαφ πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό που θεωρεί βασική της λειτουργία ε, η βασική λειτουργία της Όλαφ λοιπόν είναι το ερευνητικό έργο. Το δικαστήριο έχει δύο δείκτες για προς αυτό το σκοπό. Πρώτο απ' όλα το ποσοστό του προσωπικού που ασχολείται με ερευνητικό έργο. Δεύτερον, και επιχειρήσεις. Δεύτερον, αναλύεται ο χρόνος που δαπανάται για την ανάλυση περιπτώσεων όσον αφορά την γραφή αυτού του χρόνου που αναλύσκεται στο σύστημα της Όλαφ που εισήχθη το 2007. Παρά λοιπόν την αύξηση του προσωπικού κατά 120 άτομα από το 2005, το ποσοστό στις διευθύνσεις Α και Β παραμένει στο 40%. Η αρχική σύσταση του δικαστηρίου ζητεί σε μια ενίσχυση του ποσοστού του προσωπικού που ασχολούνται σε αυτές τις διευθύνσεις που ασχολούνται με τις επιχειρήσεις και τις έρευνες. Αυτό θα ήταν σημαντικό μέτρο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ταχύτητας και της διάρκειας των ερευνών. Το δικαστήριο επίσης στην έκθεση του καλεί την Όλαφ να εξασφαλίσει η μονάδα στρατηγικής παρακολούθησης να συμβάλλει στους στόχους της Όλαφ της προστασίας δηλαδή των συμφερόντων της Ένωσης με την διεξαγωγή ερευνών. Δεύτερο θέμα. Πρέπει να βελτιωθούν οι αναφορές και οι έρευνες Δηλαδή η αρχική έκθεση του δικαστηρίου είχε αναφερθεί σε διάφορους τομείς που μπορούσαν να βελτιώσουν αυτούς τους δύο παράγοντες. Το ένα θέμα είχε σχέση με τη διάρκεια των υποθέσεων και την γενική διοίκηση ώστε να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ξεκινώντας με την απονομή προτεραιοτήτων στις διάφορες υποθέσεις, τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, την τον καλύτερο προγραμματισμό και την συνεχή παρακολούθηση. Πρέπει να είμαστε ειδικοί και πρέπει να πούμε ότι ορισμένα μέτρα ε, υιοθετήθηκαν για να αντιμετωπιστούν ε, αυτά τα θέματα. Έχουν αναπτυχθεί ζητήματα διαχείρισης του χρόνου, έχουμε τον κανόνα de minimis, έχουμε διαδικασίες που άλλαξαν και συμφωνίες σαν για την ενίσχυση της συνεργασίας όπως αναφέρατε κυρία Πρόεδρε. Παρόλες όμως αυτές τις βελτιώσεις θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι έχει παραμείνει η διάρκεια των υποθέσεων σταθερή παρόλα αυτά και γι' αυτό το δικαστήριο θέλει να παρατρύνει την Όλαφ ώστε τα διάφορα μέτρα που λαμβάνουν να ανασκοπιστούν ώστε να εξασφαλίσουμε πρόοδο σε αυτόν το δίκτυ της ταχύτητας. Επίσης καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρα να λάβουν υπόψη τους αυτές τις ανάγκες, τις διάφορες αναθεωρήσεις σε σχέση με την Όλαφ. Έχουμε βελτίωση στις αναφορές της Όλαφ και το δικαστήριο ζητά επικέντρωση στους στόχους όπως έχουν σχεδιαστεί. Τέλος. Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η Εποπτική Επιτροπή έχει σημαντικό ρόλο να παίξει μία απόφαση το 2008 αποσαφήνισε ότι σημαντικό έργο της Εποπτικής Επιτροπής είναι να προστατεύσει τα συμφέροντα όσων υπά... υπάγονται σε έρευνα. Και έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή το εγχειρίδιο λειτουργίας της Όλαφ περιέχει οδηγίες σε σχέση με αυτό το θέμα. Η σύστασή μας λοιπόν είναι να συμπληρώσουμε τις νέες ρυθμίσεις προσδιορίζοντας μια επίσημη διαδικασία για περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εποπτική Επιτροπή θέλει να γνωμοδοτήσει για συγκεκριμένες υποθέσεις. Μια δεσμευτική διαδικασία θα βοηθήσει τη διαφάνεια και θα εξασφαλίσει η Εποπτική Επιτροπή να μην παρεμβαίνει στις έρευνες που βρίσκονται υπό εξέλιξη. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι η έκθεση του δικαστηρίου επιβεβαιώνει την ανάγκη για αναθεώρηση του κανονισμού Όλαφ δεχόμαθα ότι ε, η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία της Όλαφ πρέπει να βελτιωθούν και ελπίζουμε ότι η έκθεση βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, επεξεργαζόμαστε και μια γνωμοδότηση σε σχέση με τις αναμενόμενες ε, αναμενόμενους κανονισμούς για τη ρύθμιση της Όλαφ και ελπίζουμε ότι αυτές οι γνωμοδοτήσεις θα βοηθήσουν και αυτές προς την ίδια κατεύθυνση. Θα ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε ότι η συνεργασία με την Όλεφ κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου ήταν καλή, επικοδομητική και εκ μέρου των ελεγκτών μας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μας. Η επαφή ήταν επικοδομητική με τον νέο Γενικό Διευθυντή της Όλαφ. Είχαμε ανταλλαγή απόψεων και με την Εποπτική Επιτροπή και όλα αυτά, αν θέλετε, αποκτούν μεγαλύτερη σπουδαιότητα μέσα στο πλαίσιο της αναμενόμενης αναθεώρησης όλα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ για τα σχόλιά σας. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους βουλευτές που το ζήτησαν. Ο κύριος Μπόσιτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο και τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά. Η ειδική έκθεση λέει ότι οι στόχοι και ο σχεδιασμός είναι οι μεγάλες αδυναμίες στην έρευνα. Και δεν υπάρχει και ανεξάρτητος έλεγχος επί των ερευνών. Ούτε και διατάξεις ώστε να είναι υποχρεωμένες οι έρευνες αυτές να ακολουθούν συγκεκριμένο σχέδιο. Τα αναφέρω, τα ξανά αυτά γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι και η ουσία του προβλήματος. Έξι χρόνια μετά την πρώτη έκθεση του 2005 ε, βλέπουμε τα ίδια σχόλια. Δηλαδή ότι οι έρευνες δεν είναι παρκής, ε, δεν γίνεται αποτελεσματική κατανομή στόχων η συλλογή πληροφοριών δεν είναι αρκετή, υπάρχει έλλειψη συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Ακόμη η Εποπτική Επιτροπή δεν υλοποιεί πλήρως το ρόλο της κτλ. Αναφέρονται πολλά τέτοια σχόλια. Όταν λοιπόν μιλούμε για την αξιολόγηση Πρέπει να πούμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο έκανε πολλή δουλειά ακόμη. Πρέπει να πούμε ότι η Όλαφ έκανε πολλές προσπάθειες για να μειώσει τις αδυναμίες της. Όμως η κατάσταση είναι όπως είναι. Λοιπόν, τίθεται συνεπώς το ερώτημα, τι θα γίνει στη συνέχεια. Γιατί δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τον έλεγχο και τα ένομα μέσα που χρειαζόμαστε. Έχουμε μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, έχουμε 27 κράτη-μέλη σήμερα, ίσως και περισσότερα στο μέλλον. Συνεπώς έχουμε μεγαλύτερο έργο προς πραγματοποίηση και οι νομικές πράξεις είναι περισσότερες, αυτές που πρέπει να συνταχθούν δηλαδή, και όλα αυτά πρέπει να προσαρμοστούν χωρίς οι διαδικασίες δηλαδή πρέπει να προσαρμοστούν χωρίς να υπάρξει επέκταση. Πρέπει να καταργηθούν ουσιαστικά οι λόγοι για τους οποίους καθυστερεί η εργασία καθημερινά. Διαπιστώνεται μια έλλειψη συλλογής στοιχείων επίσης. Επανειλημμένα έχω πει ότι η συλλογή στοιχείων στα κράτη-μέλη είναι σημαντική τα στοιχεία αυτά πρέπει να δίδονται στην Όλαφ και η Όλαφ πρέπει να είναι περισσότερο ενεργή προς αυτή την κατεύθυνση και εμείς πρέπει να στηρίξουμε την Όλαφ σε αυτές τις προσπάθειες. Ε, δηλαδή θα νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε από την Κομισιόν ε, να επιβάλλει ορισμένες αρχές στις δημόσιες προμήθειες ώστε όταν χρησιμοποιούνται δημόσια κονδύλια να εφαρμόζονται οι αξίες οι σωστές για τις δημόσιες προμήθειες. Έχουν πραγματοποιηθεί πρόοδοι σε πολλά κράτη-μέλη, αλλά τα συστήματα δεν χρησιμοποιούνται ευρέω, τα σωστά συστήματα δεν χρησιμοποιούνται ευρέω, διότι δεν υπάρχει πολιτικό ενδιαφέρον γι' αυτό. Συνεπώς, μελλοντικά, θα πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτια και να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε το έργο και για την Όλαφ και για το ελεγκτικό συνέδριο και για την ε, Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Τώρα λοιπόν ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γιάλα Σέντα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά κύριε Πρόεδρε και ως συγγητή για το ενδιαφέρον έγγραφο εργασία και να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκαλέα, το αρμόδιο μέρος του Ελεκτικού Συνεδρίου για την ειδική έκθεση. Η έκθεση αυτή αφενός επισημαίνει μια σειρά ελλείψεων και αδυναμιών που φυσικά μας ανησυχούν, τα μάλα, γιατί δείχνουν ότι ένας τόσο σημαντικός οργανισμός όπως είναι η Όλαφ που θα πρέπει να το έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί ασχολείται με την καταπολέμηση απάτη και θα πρέπει να έχει αυτονόητη αξιοπιστία, βλέπουμε ότι η ΟΛΑΦ δεν ακολούθησε όλες τις συστάσεις ε, από την πρώτη δική έκθεση, ούτε έχει βελτιωθεί αισθητά στα θεμελιώδη στοιχεία που αυτές επισημαίνουν. Αυτό με ανησυχεί. Γιατί η σύσταση του να επικεντρώνεται κυρίως η ΟΛΑΦ στις έρευνες δεν έχει εφαρμοστεί. Επισημαίνουμε εδώ ότι χωλαίνει ακόμη η κατάσταση στην ΟΛΑΦ και ελπίζω ο νέος διευθυντής να λάβει υπόψη αυτό το πρόβλημα και να διορθώσει την κατάσταση. Γιατί αφιερώνουμε πολλούς πόρους σε αυτό το θέμα και το θέμα της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των στοιχείων. Θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε η μοναδική δυνατότητα που έχει η ΟΛΑΦ για έρευνες να μην πάει χαμένη. Θα πρέπει ταυτόχρονα να δίνονται και όλα τα εχέγγυα. Γιατί εγώ από την αρχή του έργου μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέτησα ένα διοντολογικό κώδικα που να εξασφαλίζει όλες αυτές τις εγγύσεις. Γιατί σε πολλές υποθέσεις έχουμε τέτοια φαινόμενα. Δεν δίνονται απαραίτητα εχέγγυα, κάτι που αποβαίνει εις βάρος τη ε, της ΟΛΑ. Φαίνεται ότι δεν δίνονται εχέγγυα τήρηση των δικαιωμάτων των ε, ανθρώπων που υπόκεινται σε έρευνε. Θα πρέπει αυτά τα εχέγγυα να είναι εξασφαλισμένα και τα δικονομικά. Γιατί είδαμε υποθέσει, είδαμε περιπτώσει όπου έκανε κάθεση Όλαφ. Και μάλιστα μετά από δύο χρόνια τα ατασταλιών είδαμε ότι και στα δικαστήρια δημιουργήθηκε πρόβλημα για την ΟΛΑΦ γιατί μετά από πολύχρονες έρευνες και κατηγορίες της ΟΛΑΦ για τους ε, υπόπτους τελικά θώνονταν από το δικαστήριο παρόλο που είχαν καταστρατηγηθεί σημαντικά δικαιώματα και εγγύης τους. Το χειρίδιο κατά τη γνώμη μου δεν αρκεί. Αν δεν υπάρχει κάποιος ε, δεοντολογικός κώδικας, τουλάχιστον υπάρχει μια επιτροπή επαγρύπνησης. Ε, να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των ερευνών, αλλά δεν σημαίνει η ε, ανεξαρτησία των ερευνών ότι ο ΛΑΦ γίνεται ένας οργανισμός που ξεφεύγει από τον έλεγχο και μπορεί να υπονομεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των ενδιαφερομένων. Και το θέμα της παράτασης των προθεσμιών είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε ένα εξυγχρονισμό των συστημάτων, είχαμε μια αύξηση των πόρων. Γιατί λοιπόν συνεχίζεται αυτή η κολυσιεργία και αυτή η χρονοτριβή σε ό,τι αφορά την διερεύνηση ορισμένων υποθέσεων που μερικές κρατάνε χρόνια ολόκληρα, κάπου υπάρχουν σκόπελοι που εμποδίζουν την ε, διεξαγωγή των ερευνών. Υπάρχουν ίσως και άλλες αιτίε πέραν της ανεξαρτησίας του ελέγχου και των ερευνών. Ο κύριος Γκαλέα λοιπόν, που εντόπισε κάποιες δυσκολίες και αδυναμίες αυτού του σημαντικού οργανισμού που είναι η ΟΛΑΦ, υπέβαλε κάποιες ε, συστάσεις και ευχαριστώ και τον εισηγητή μας, τον κύριο Ντόιτς, που στη δική του έκθεση τη εστερνίζεται και μπορούμε να βοηθήσουμε και εμεί ω Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού την ΟΛΑΒ για να βελτιώσει το συντομότερο δυνατό την κατάσταση αυτή. Και ελπίζω στο πρόγραμμα εργασιών που θα μα υποβάλει ο νέο διευθυντή τη ε, να βελτιωθεί η διαχείριση και να βελτιωθεί και η συνεργασία με τη Eurojust ώστε να δημιουργηθεί ένα διαφανές και αξιόπιστο πλαίσιο ελέγχου για τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί η ΟΛΑΦ είναι απαραίτητη για τους πολίτες, αλλά θα πρέπει να είναι σωστά πλαισιωμένη για να αποφευχθούν οποιοδήποτε είδους παρεκτροπές. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ε, και εγώ την έκθεση ε, του Ελεγκτικού Συνεδρίου τη βρίσκω πολύ καλή και η έκθεση δείχνει ότι κάλλιστα μπορεί κανείς ε, να εκφράζεται με αριθμούς και οποτεδήποτε κανείς εκφράζεται με αριθμούς ε, γίνεται και κατανοητός. Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Ε, λοιπόν, συγκεκριμένα, πόσους ανθρώπους χρησιμοποίησε η Όλαφ για την ουσιαστική ερευνητική δραστηριότητα, το ελεγκτικό συνέδριο λέει περίπου το 37% και η Επιτροπή απαντάει στο πίσω μέρος ότι το ποσοστό είναι 75% και ο Γενικός Διευθυντής ε, όταν μίλησε είπε ότι και εκείνος και οι άλλοι ε, θα θελήσουν να φτάσουν το 50%. Γι' αυτό ερωτώ, ο αριθμός ε, εκείνων που ασχολούνται αυτή τη στιγμή με τις έρευνες, ποιο είναι το ποσοστό τους? Πολύ ωραία. Το λόγο έχει ο κύριος Μικελάτ που εκπροσωπεί την Όλαφ και μπορεί να λάβει το λόγο στη σύντηση μας με αυτή του την ιδιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Τζοβάνι Κέσε, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα γιατί είχε εδώ και πολύ καιρό ηλυμένες υποχρώσεις στην Παγκόσμια Τράπεζα και στα Ηνωμένα Έθνη. Βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική σε διάφορες ε, πολιτείες και δεν, μπορεί, δεν θα μπορούσε να είναι εδώ. Πάντως ε, ήταν ε, στις Βρυξέλλες εδώ και δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Το είδα με τα μάτια μου αυτό. Δούλεψε ολόκληρα Σαββατοκύριακα και τις νύχτες και πραγματικά λυπάται πάρα πολύ που τελικά σήμερα ειδικά δεν μπόρεσε να έρθει να μιλήσει για ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί στην υπηρεσία μας από τότε που διορίστηκε ο ίδιος. Εγώ λοιπόν ομιλώ τόσο εκ μέρους της Επιτροπής όσο και εκ μέρους της ε, Όλαφ. Αν χρειαζόταν ε, να ε, κάνω διάκριση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ρόλους θα το έκανα και θα το κάνω αν χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για, όλα, για αυτά τα χρήσιμα σχόλια που κάνατε και για τις συστάσεις σας. Ξέρω ότι ο κύριος Κέσλε θα λάβει σοβαρά υπόψη του τις συστάσεις αυτές στα σχέδιά του της αναδιάρθρωσης, κυρίως όταν θα επιληφθεί όλο αυτό το οικοδομήματος που φέρει τον τίτλο ερευνητική διαδικασία. Και αυτό θα σας το εξηγήσω με περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα. Πριν λοιπόν αναφερθώ σε αυτήν την έκθεση, θα μου επιτρέψετε ίσως να σχολιάσω και κάποια πράγματα που ελέγχθησαν στην προηγούμενη έκθεση, που ε, είναι παλιά έξι ετών. Βεβαίω εδώ τίθεται το ερώτημα κατά πόσον ε, ε, το ποτήρι είναι ε, ποσοστά, είναι γεμάτο ή άδειο με κατά τρίτον, 15, 8, 3 5 Γιατί ξέρετε τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι εμείς έχουμε εφαρμόσει τις συστάσεις σα βέβαια σε διαφορετικό βαθμό και θα δείτε ότι Όσον αφορά τις συστάσεις στη νέα έκθεση, εκεί δεν δεχτήκαμε πλήρης και αυτούσιες όλες τις προτάσεις σας, γιατί κρίναμε ότι τα πράγματα αλλάζουν και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να αλλάξει και η δική μας συστάση σε σχέση με ορισμένα θέματα. Ας επανέλθουμε τώρα στην παρούσα έκθεση. Εμείς σε γενικές γραμμές ε, συμφωνούμε με το αποτέλεσμα. Βεβαίω ε, η Επιτροπή στην απάντησή της ε, ανέφερε με πολλές λεπτομέρειες τις απόψεις της και εμείς όσο Όλαφ συμβάλαμε σημαντικά σε αυτή την τοποθέτηση της Επιτροπής. Από το 2005 λαμβάνεται υπόψη αυτή η διαδικασία. Είναι αλήθεια ότι η διαδικασία έχει παραμείνει σταθερή, δεν έχει αλλάξει. Εμείς από τη δική μας την εμπειρία μπορούμε να σας πούμε ότι σε γενικές γραμμές οι υποθέσεις έχουν γίνει πιο σοβαρές και πιο περίπλοκες. Τα τελευταία στοιχεία από το 2010 καταδεικνύουν μία μικρή μείωση στην διάρκεια των ερευνών από κάτι πάνω από δύο χρόνια σε κάτι λιγότερο από δύο χρόνια. Έχουμε επίσης ε, καταρτήσει μία προσέγγιση de minimis, η οποία μας επιτρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε πιο περίπλοκες υποθέσεις. Εξάλλου, έχουμε ενισχύσει ε, τις ε, πληροφορίες στρατηγικής σημασίας που συλλέγουμε. Το ε, βέβαια δεν είναι πάντα εύκολο γιατί δεν είναι ε, σε αρμονία με τις ε, αποφάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου το οποίο πρέπει να έχει αποχρόντες λόγους για να επιτρέψει αυτές τις στρατηγικές πληροφορίες. Αυτές οι στρατηγικές πληροφορίες είναι σημαντικότερες για την πρόληψη απάτης και η Επιτροπή θεωρεί ότι και αυτό είναι μια πολύ σημαντική πράξη, γι' αυτό λοιπόν θα συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν χρειάζεται νομίζω να σας πω, ιδιαίτερα σε εσά κύριε Πρόεδρε, ότι η νομοθετική διαδικασία αυτή τη στιγμή θα δώσει τη δυνατότητα στους θεσμούς να ε, αντιμετωπίσουν τα θέματα που τους αφορούν μόνοι τους το 2005 υπάρχει μια έκθεση και αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και να ληφθεί υπόψη μόνο εφόσον υπάρξουν αλλαγέ ε, στη νομοθεσία. Όπω σα είπα λοιπόν, δεχτήκαμε εν μέρη ή πλήρωση τι συστάσει. Ε, καταβάλαμε κάθε δυνατότητα για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των ερευνών μα. Όσον αφορά Στη διάρκεια, σας είπα, προσπαθούμε να τη μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Βεβαίω, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια πολύ περίπλοκη δοκιμή, ε, δομή ε, και δικαστική και άλλη μορφή που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που θα επιθυμούσαμε. Ε, ο κύριος Κέσλα... Όσον αφορά τις συστάσεις προσβλέπει σε μια εσωτερική αναδιοργάνωση που θα επιτρέψει την εφαρμογή των συστάσεων αυτών και νομίζω ανέφερε και στην επιστολή του κύριε Πρόεδρε, στην επιστολή που σας έστειλε την Παρασκευή, ότι προσβλέπει στο να συζητήσει μαζί σας το θέμα αυτό, οποτεδήποτε βέβαια η Επιτροπή σας κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Χωρίς να θέλω βέβαια να προκαταβάλω ε, τις αποφάσεις του. Ε, θέλω μόνο να σας πω ότι τα σχέδιά του καλύπτουν την λειτουργική αποτελεσματικότητα, ε, τον εξορθολογισμό, την πιο εξορθολογισμένη δομή των ερευνών, μικρότερη διάρκεια και επίσης και περαιτέρω χρήση της προσέγγισης de minimis. Όσον αφορά τώρα στο θέμα του προσωπικού, το ποσοστό του προσωπικού που απασχολείται με έρευνες. Όπως όλα τα στατιστικής φύσεως θέματα, καταρχήν είναι θέμα ορισμού. Η προσέγγιση που χρησιμοποιεί το ελεγκτικό συνέδριο είναι η εξής, ε, να υπολογίζει κανείς ε, τους ανθρώπους ε, ε, τις κατηγορίες Α και Β. Αυτό όμω δεν αφορά όλους όσοι εμπλέκονται στην έρευνα. Παραδείγματο χάρη, μια ερευνητική ομάδα που κάνει μια επιτόπια έρευνα ε, χρησιμοποιεί αναλυτές ε, υπολογιστών. Αυτή δεν είναι πάλι Α ή Β ή χρησιμοποιεί και άλλο προσωπικό που δεν ανήκουν στην Γενική Διευθυνσία Α ή Β η ομάδα που ε, στηρίζει την, τις έρευνες ε, να ε, συντάσσεται ο φάκελος να συλλέγονται πληροφορίες και αυτοί δεν ανήκουν στην Γενική Διεύθυνση Α ή Β. Άρα δηλαδή καταλήγουμε στο ότι η προσπάθειά μας, αν λάβει κανείς υπόψη του και την άλλη πλευρά, μπορούμε να μιλάμε για ένα περίπου 75% του προσωπικού. έτσι απορρέει έτσι προκύπτει αυτό το ποσοστό. Αν δείτε τώρα και τον αριθμό των υπαλλήλων οι οποίοι είναι μόνο ερευνητές, τότε το ποσοστό μειώνεται σε λιγότερο από το ίμιση. Και θεωρώ ότι αυτό το, ποσοστό πρέπει εσείς να συγκρατήσετε, το 50%. Όμως, ε, όπως σας είπα, το σύνολο του προσωπικού που ασχολείται με τις έρευνες και με συντονισμό, σας είπα ότι αυτό αντιστοιχεί στο 75%. Ένα άλλο στοιχείο, ένας αριθμός που αναφέρθηκε σήμερα είναι το 37% του χρόνου που δαπανάται για έρευνες ε, και πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά το ποσοστό αυτό έχουμε κάποιο πρόβλημα, βέβαια από εμά προκύπτει, εμείς δεν νομίζουμε ότι σωστά αναφέρεται ο χρόνος. Γιατί σχεδόν όλοι οι ερευνητές δεν έχουν ε, καμία λερμοδιότητα πέρα από την έρευνα. Ίσως να δαπανάνε κάποιο χρόνο στη διοίκηση. Αυτό συμβαίνει όταν καλούνται να συντάξουν μία έκθεση ή ε, όταν ε, κάνουν ερωτήσεις στον ύποπτο που θέλουν να εξετάσουν. Υπάρχουν λοιπόν αντιφάσεις όσον αφορά αυτό το ποσοστό. Και αυτό το ερευνά ο κύριος Κέσε. Θα τα λάβει όλα αυτά υπόψη του στις αποφάσεις που θα λάβει. Όσον αφορά τώρα την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των εγγυήσεων, βεβαίως ε, μας ε, ελέγχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όλο και περισσότερο Και αυτό είναι κάτι που θα ληφθεί υπόψη στην συνεχιζόμενη νομοθετική διαδικασία. Νομίζω ότι καλύτερα να μιλήσουν άλλοι για το μέλλον, καλύτερα από μένα. Και το τελευταίο που θέλω να θίξω είναι ότι προσπαθούμε με διάφορους τρόπους ε, να ε, βελτιώσουμε τη συνεργασία μας ε, με τα κράτη-μέλη και με τη Eurojust. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να εξελιχθεί, να προκύψει από μόνο του. Δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Πάντως ε, προσβλέπουμε και σε αυτόν τον τομέα σε περαιτέρω βελτίωση κατά τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ για αυτά τα πολύ αξιόλογα σχόλια. Ε, τελειώνει ο χρόνος μας έπρεπε να έχει ξεκινήσει η συνάντηση των συντονιστών πριν από 15 λεπτά ήδη. Το θέμα όμως είναι σημαντικό, όχι μόνο επειδή είμαι υπεύθυνο για αυτό το φάσμα, αλλά πιστεύω ότι το θέμα είναι πραγματικά περσέ σημαντικό, από μόνο του. Με την άδειά σας λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Εποπτικής Επιτροπής της Όλαφ και μετά θα δώσω δύο λεπτά στον κύριο Γκαλέα για να σχολιάσει όσα άκουσε σήμερα. Δεν θα συνοψίσω προσωπικά όσα ακούσουμε. Εγκαταλείπω το δικαίωμά μου <laughs> αυτό. Λοιπόν, ποιος θα μιλήσει εκ μέρους της Εποπτικής Επιτροπής, παρακαλώ. Βλέπω διάφορους εκπροσώπους. Ένας από εσά μπορεί να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε στην Επιτροπή σας. Είμαστε δύο μέλη της ε, Εποπτικής Αρχής ε, της Όλαφ. Η συνάδελφός μου, Ρόσελιν Ράιτ και εγώ που προεδρεύω σε αυτή την Επιτροπή. Ε, είχαμε λοιπόν στενές επαφές με το ελεγκτικό συνέδριο για να συζητήσουμε για την έκθεση αυτή και θέλω να σας πω ότι αυτά τα οποία ακούσαμε μέχρι τώρα είναι εκείνα τα οποία και εμείς έχουμε συμπεράνει ως ε, Επιτροπή Εποπτείας. Και φαντάζομαι ότι τις γνωμοδοτήσεις που σας ε, αποστέλουμε, γιατί σας στέλνουμε πάρα πολλές κάθε χρόνο, τις διαβάζετε και νομίζω από αυτές ε, μπορείτε να συνάγετε ότι εμείς ε, επιθυμούμε να ασκούμε έλεγχο. Αυτό είναι το βασικό και με βάση αυτό συντάσσουμε τις εκθέσεις μας. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, που είναι συνέχεια των προηγούμενων εκθέσεων, κυρίως αυτής του 2005, τα θέματα είναι λίγο πολύ τα ίδια. Και εσείς το είπατε αυτό. Παρότι βέβαια, εντωμεταξύ, έχουν περάσει πέντε χρόνια Τίθεται βέβαια το ερώτημα κατά πόσον η νομική βάση που διέπει την Όλαφ εξακολουθεί να ισχύει όχι. Όχι λοιπόν, πρέπει να τροποποιηθεί. Και κατόπιν τούτου η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. Θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα σε τρία σημεία, όπου το ένα βέβαια θα τον αλάβει η κυρία Ρόσελιν Ράιτ. Το πρώτο που θα πω εγώ αφορά την ε, συγκέντρωση αρμοντήτων της Όλαφ. Πρόκειται για την έρευνα και έρευνα και εποπτεία σε οποιαδήποτε ερευνητική δραστηριότητα διεξάγεται. Κατόπιν, βελτίωση των αποτελεσμάτων μέσα από καλύτερο προγραμματισμό. Ε, σε αυτό θα τοποθετηθεί η κυρία Ράιτ. Πρώτο θέμα, συγκέντρωση στην βασική ε, δραστηριότητα. Νομίζω ότι από αυτού δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά. Ήδη έχουν αναφερθεί αριθμοί, όμως ε, νομίζω ότι αυτό το θέμα, το θέμα της ε, βασικής ε, δραστηριότητας, όπως ακριβώς ελέγχθη και τέθη από εμάς, κύριε Άλεν Τενέβη καταφατικά το ξέρετε, εδώ λοιπόν δεν πρέπει να δίνουμε σημασία μόνο στους αριθμούς, αλλά χρειαζόμαστε και ορισμό του όρου έρευνα. Τι είναι η έρευνα? Έρευνα μεταξύ άλλων είναι συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών. Και αυτό είναι έρευνα. Κατόπιν τούτου, το ποσοστό που αναφέρεται για ε, τις διευθύνσεις Α και Β δεν είναι απόλυτα σωστό και το ποσοστό είναι πολύ χαμηλό σε σχέση και με άλλα κατοίκοντα που ε, εκπληρώνονται χωρίς όμως να είναι άμεσα αρμοδιότητα της Όλαφ γιατί η Όλαφ είναι ένας φορέας ο οποίος ε, καλείται να διεξάγει διοικητικές έρευνας προς όφελος των συμφερόντων για να προστατεύσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο ρόλος της Όλαφ. Το 50% λοιπόν των ε, συνεργατών μας, του προσωπικού μας, χρησιμοποιείται για έρευνες. Εγώ ήδη παλαιότερα ε, σας είπα ότι θα προσπαθήσουμε να αυτό μας το στόχο. Το ελεγκτικό συνέδριο πολύ σωστά είπε ότι η διάρκεια ερευνών δεν μειώθηκε σημαντικά. Ξεκολουθούμε να έχουμε μεγάλα χρονικά διαστήματα ερευνών, κατά μέσο όρο 25 μήνες. Και ο 7,1 μήνες, 7 μήνες περίπου ε, ε, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση. Σωστά ελέγχθη ότι αυτά τα διαστήματα είναι μακριά, είναι μεγάλη η διάρκεια των ερευνών. Και αν δεν περιοριστεί η διάρκεια των ερευνών, τότε πρέπει να ξαναδούμε τι έρευνες πρέπει να λαμβάνει η Όλαφ. Οι υποθέσεις τώρα είναι πολύ πιο περίπλοκες. Άρα δηλαδή ε, Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός του προσωπικού που ασχολείται με τις έρευνες. Το έχουμε συζητήσει αυτό επανειλημμένα με το ελεγκτικό συνέδριο. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να αλλάξουμε και τον τρόπο εργασίας και τη δομή της Όλαφ. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε αλλαγές απλά μετακινώντας οργανογράμματα και μεταθέτοντας ε, υπαλλήλους. Πρέπει να υπάρξουν σαφείς αποφάσεις και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Όλαφ και χρειάζονται και συνοδευτικά μέτρα και μέτρα περαιτέρω κατάρτισης. Η ε, Επιτροπή Εποπτείας θα δώσει ιδιαίτερη σημασία ε, στο θέμα αυτό. Κάτι άλλο οι κύριοι βουλευτές είπαν με απόλυτη σαφήνεια ότι το θέμα του ελέγχου της Όλαφ ε, δεν εκφράστηκε με απόλυτη σαφήνεια. Και αυτό το είπε και το ελεγκτικό συνέδριο, ότι δεν έχει διασφαλιστεί ακόμα η αμεροληψία των ελέγχων, η απόλυτη ανεξαρτησία τους. Κατόπιν τούτου πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές έτσι ώστε να απλουστευτούν λιγάκι οι νομοθετικές διατάξεις γιατί νομίζω αυτό το επιδιώκει και η Επιτροπή σας αν έχω καταλάβει καλά. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε στο νομοθέτη ε, μία πρόταση για τροποποίηση της οδηγίας 1073 του 99 και θεωρώ ότι ε, λαμβάνονται υπόψη κάποια αιτήματά μας, όχι όμως όλα τα σημεία του σχετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ήδη το 2008 υιοθέτησε το ψήφισμα αυτό. Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας ε, ε, τις οποίες προβάλλει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτές οι αρμοδιότητες ε, και κυρίως όσον αφορά τον έλεγχο των διαδικασιών θα πρέπει να επεκταθούν και εκτός αυτού θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Όλαφ και των τριών διαφορετικών οργάνων. Είμαι πεπισμένη ότι η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ε, Όλαφ είναι απολύτως απαραίτητη εφόσον επιθυμούμε αποτελεσματικότητα και ε, ανεξαρτησία ελέγχων. Η Επιτροπή Υποπτίας είναι εκείνη που κατά κύριο λόγο μπορεί να διασφαλίσει τη σωστή διάρκεια των ερευνών και ο έλεγχος ε, αυτός δεν θα πρέπει βεβαίως ε, να γίνεται παντελώς αποκομμένος. Ο έλεγχος ε, θα πρέπει να, απο... να δίδει και κάποιες ε, πληροφορίες ενδιαφερόμενους. Εξάλλου, η Επιτροπή Εποπτείας δεν προτίθεται και δεν φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το Γενικό Διευθυντή, ούτε θέλει να παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια των ερευνών μέσα από το διάλογο, είτε μέσα από την τροποποιημένη πρόταση της Κομισιόν, είτε μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα από την διαδικασία που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου θα καλείται και η Επιτροπή Υποπτίας μέσα από αυτό επιθυμούν τα διάφορα όργανα να ε, καταλήξουν στο ότι η Όλαφ εργάζεται σωστά. Γιατί στη τελική ανάλυση η Επιτροπή Εποπτείας είναι εκείνη που κατά κύριο λόγο μπορεί να σας προσφέρει αυτή τη βεβαιότητα. Για να επιτευχθεί όμως ο στόχος η Επιτροπή Εποπτείας ε, πρέπει να ορίζεται ο όρος επιτροπής αυτής στον κανονισμό και επίσης η επιτροπή αυτή να έχει τα, το νομικό και εξοπλισμό και το απαραίτητο προσωπικό για να μπορεί να διεξάγει τον απαραίτητο έλεγχο. Ε, και στην περίπτωση αυτή τα δικαιώματα των φυσικών και των νομικών προσώπων προφανώς και προστατεύονται. Τέτοιου είδους έλεγχος θα συνέβαλε επίσης ε, στο η νομολογία πρώτης βαθμίδας ε, δικαστηρίων ε, να τηρούνται τα δικαιώματα αυτά, να προστατεύονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Eh, eh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ράιτ και να τη θέλω να παρακαλέσω να μην ξεπεράσει το δίλεπτο αν γίνεται, γιατί έχουμε καθυστερήσει πολύ και οι συντονιστές θα δυσαρεστηθούν. Θα μου κόψει το κεφάλι αν δεν ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνική. Εμένα τους τελευταίους μήνες με απασχόλησε κυρίως ο έλεγχος και η διαχείριση των ερευνών στην ΟΛΑΦ. Και αυτό αφορά όσα είπε η ΟΛΑΦ για τη διάρκεια των ερευνών και την αποτελεσματικότητα του λειτουργικού ρόλου της ΟΛΑΦ. Και φυσικά ένα από τα στοιχεία είναι η αποτελεσματική ο αποτελεσματικός σχεδιασμός των ερευνών και η παρακολούθηση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ε, εντός των μονάδων της ΟΛΑΦ. Γι' αυτό και η Συμβουλευτική Επιτροπή μας έχει συντάξει σχετική γνωμοδότηση και χαίρομαι γιατί ήδη διαπιστώσαμε κάποια πρόοδο και μάλιστα μια ε, αρμόδια Γενική Διεύθυνση εφαρμόζει ήδη τις προτάσεις μας και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα διαπιστώσουμε συντόμευση της διάρκειας των ερευνών, κάτι που είναι ζωτική σημασία, εξαιτία του αποτελεσματικότερου σχεδιασμού των ερευνών και της, του αυστηρού ελέγχου της διαχείρισης από την ίδια την ΟΛΑΦ. Και εκεί η Συμβουλευτική Επιτροπή θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. Φυσικά εμείς δεν μπορούμε να παρεύουμε σε τρέχουσες έρευνες και αυτό περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις ελεκτικές μας αρμοδιότητες, αλλά σίγουρα θα παρακολουθούμε άγρυπνα την εφαρμογή των συστάσεών μας. Και νομίζω ότι χάρη στην εφαρμογή τους και θα βελτιωθούν οι έρευνες, η αποτελεσματικότητά τους, αλλά και θα συντομευθεί η διάρκεια, η διάρκειά τους, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που ήσασταν τόσο λακωνική μεν, αλλά ε, περιεκτική δε. Και για δύο λεπτά, πριν ολοκληρώσω τη συνεδρίαση, ο κύριος Γκαλέα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα τρία μέλη της Επιτροπής που έχουν λάβει το λόγο σήμερα ε, έχουν θίξει θέματα τα οποία συνεχίζουν να είναι μεγάλο ενδιαφέροντος για αυτή τη συζήτηση και για αυτόν τον τομέα, τον συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι η έκθεση του δικαστηρίου αντιμετωπίζει σε λεπτομέρεια και σωστά τα θέματα που έθιξε η κυρία Γκρέσλερ όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την διαχείριση των επιχειρήσεων Όλαφ. Ο κύριος Άλεφ επίσης έδωσε τη θέση της Όλαφ πάνω σε αυτό το θέμα. Το άλλο ζήτημα που κατά την άποψή μου είναι πολύ σπουδαίο είναι αυτό που ετέθη από την κυρία Άιλα Σέντερ όσον αφορά την επαγρύπνηση της Όλαφ και των επιχειρήσεων. Το δικαστήριο πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θα επαρκούσε για να πραγματοποιήσει αυτή την παρακολούθηση, εποπτεία. Πιστεύω ότι τρόπον την θα υιοθετούσαμε μια διαφυγή αν βασιζόμαστε σε αυτόν τον τύπο της εποπτείας. Χρειαζόμαστε κάτι που αφορά την καθημερινή εργασία. Κάτι που να είναι αποτελεσματικό, ώστε όλοι να είμαστε ήσυχοι ότι ο Όλαφ λειτουργεί με όλο το δυναμικό όσο καλά μπορεί, αλλά μέσα στο πλαίσιο της ένομης τάξης. Όσον αφορά το θέμα που έθιξε ο κύριος Μπαλτσίτης, νομίζω ότι το πρόβλημα εκεί δεν έχει σχέση με την Όλαφ, Είναι, αφορά το Συμβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο, την Κομισιόν. Εάν δεν λύσουμε αυτό το θέμα της διπλής αποστολής της Όλαφ, πάντοτε η Όλαφ θα βρίσκεται στριμωγμένη μεταξύ δύο λειτουργιών και το ελεκτικό συνέδριο θα συνεχίζει να κάνει κριτική ανάλυση ότι δεν επικεντρώνονται παρκώς στην ερευνητική τους εργασία που είναι ο πυρήνας της λειτουργίας τους. Ευχαριστώ. Αγαπητά μέλη, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για τη συμβολή σας. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Εποπτικής Επιτροπής, ευχαριστώ όσους συνέβαλαν σε αυτή την πάρα πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έληξε και το θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης, έληξε και η συνεδρίασή μας. Θα επανέλθουμε σε 9 το πρωί. Ε, άρχεται τώρα η συνεδρίαση των συντονιστών. Θα είμαστε πολύ σύντομοι. Προτού περάσουμε στην συνεδρίαση των συντονιστών, παρακαλώ όσοι δεν πρέπει να παραμείνουν να εξέλθουν τις αίθουσες. Ευχαριστώ.